Κυρίε και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων που είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκηρύξω την έναρξη της διάσκεψης των Προέδρων που είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον κύριο Σεύκοβιτς που είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε κάποιο διαδικαστικό θέμα. Παρακαλώ κύριε Άλβαρο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μπορούσατε ενημερωτικά να μας εξηγήσετε γιατί επιλέξατε αυτό το βήμα της διάσκεψης των Προέδρων για τη συζήτηση με τον κύριο Φανερόμπο, γιατί συνήθως ε, στην Ολομέλεια γίνεται μια έκτακτη συνεδρίαση για να μπορεί να είναι για όλα τους ευρωβουλευτές. Μπορείτε να μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτή τη μορφή σήμερα. Επιλέξαμε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο για αυτή τη συνεδρίαση για να συζητήσουμε με τον πρόεδρο Πόη γιατί πρόκειται για μια συνεδρίαση που μπορεί εύκολα να συγκληθεί μετά αμέσω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή. Ε, αν θέλαμε να ακούσουμε τον κύριο Φανόμπο στην Ολομέλεια θα έπρεπε να περιμένουμε. Έγινε μια φορά που η έκθεση του κυρίου Φαν Ρομποϊ ακολούθησε τρεις εβδομάδες μετά από την ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου και θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ καιρό, γιατί εντωμεταξύ έγιναν πολλά σημαντικά γεγονότα. Θέλαμε λοιπόν να συναντηθούμε μαζί του όσο γινόταν πιο γρήγορα. Τρίτη σήμερα ε, το Συμβούλιο έλαβε χώρα την Παρασκευή. Η αίθουσα είναι ανοιχτή για όλους τους ευρωβουλευτές. Μπορούν όλοι να έρθουν και να... θέσουν ε, είτε διαδικαστικό θέμα, είτε να μιλήσουν στη διαδικασία ΚΑΣΔΙΑΙ. Εύκολα μπορεί κανείς να πάρει το λόγο. Αυτό λοιπόν έγινε προς χάρη ταχύτητας. Εγώ ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί δεν είναι παρούσα η Προεδρία, πού είναι η Ουγγρική Προεδρία, is uh, uh, as usual because it is Κοιτάξτε, είναι μια έκθεση που μας παρουσιάζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έτσι γίνεται συνήθως. Παλαιότερα, όταν η Προεδρία του Συμβουλίου μας έκανε έκθεση, όταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου μας κάνει αναφορά, δεν είναι παρούσα η Προεδρία, γιατί δεν θέλουμε να συγχαίουμε όλους ε, τους θεσμούς. Εμείς φυσικά και ε, θέλουμε να είναι και η Προεδρία παρούσα. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον, αλλά τώρα έχουμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εδώ για να μας κάνει την αναφορά του. Είναι μια τυπική διαδικασία. Ευχαριστώ. Uh, Άλλη ερώτηση, ναι, ευχαριστώ κατά την ε, προπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου για την ενέργεια και την καινοτομία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν κατάλαβα καλά την επιστολή του, έγραψε στους αρχηγούς κρατών την ίδια μέρα στις 2 Φεβρουαρίου για να προσθέσει και άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη χονδρικά την οικονομική κατάσταση. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Αλλά το Κοινοβούλιο μα δεν ενημερώθηκε για την προσθήκη αυτού του σημείου στην ημερήσια διάταξη. Διερωτώμε λοιπόν πώ εμεί μπορούμε να συζητήσουμε από πολιτική άποψη την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε την ημερήσια διάταξη που θα απασχολήσει το Συμβούλιο. Εμείς είχαμε ενημερωθεί για αυτή την αλλαγή και γενικότερα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να προτείνω ο, μήπως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μπορούσε να έρθει για να προετοιμάσουμε και την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι, καταλαβώ. Κοιτάξτε. Σταματήστε τα διαδικαστικά, γιατί έχουμε εδώ τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπροστά μα. Μπορούμε να τον ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Και έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση για όλου, για όλου του Ευρωβουλευτέ. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Σας παρακαλώ, Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να βρίσκομαι εδώ και να σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λίγες μόνο μέρες μετά τη διεξαγωγή του και όχι εβδομάδες μετά όπως συνέβη τις δύο τελευταίες φορές παρόλο που αναφέρεται στις συνθήκες και εγώ σέβομαι τις συνθήκες που οι συνθήκες λένε ότι στην Ολομέλεια γίνεται αυτή η συζήτηση κανονικά. Ευχαριστώ πάντως τους Πρόεδρους, τη διάσκεψη των Πρόεδρων που οργάνωσε την σημερινή συνάντηση εδώ λίγες μόνο μέρες όπως είπαμε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα εκείνο το οποίο βρίσκεται και στο κέντρο των σκέψεων όλων μας. Αίγυπτος. Βόρεια Αφρική. Το συζήτησε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μετά τα γεγονότα στο Κάιρο και σε άλλες Αιγυπτιακές πόλεις. Και εγκρίναμε και μια πολιτική δήλωση για την Αίγυπτο και την περιοχή. Τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό είναι κάτι που το δεχόμαστε διότι βλέπουμε ότι ο κόσμος αγωνίζεται για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη εκεί. Οι πλατείες, εκεί όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να αγωνιστούν ε, υπέρ ε, της ελευθερίας, είναι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ε, τα δικάζουμε τη βία και τον εκφοβισμό. Αυτή είναι η πολιτική μας δήλωση και θέλουμε οι επιθυμίες του Αιγυπτιακού λαού να γίνουν σεβαστές, όχι με καταστολή. Θέλουμε να υπάρξει μια ειρηνική περίοδος μετάβασης στη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως την ειρηνική αυτή μετάβαση στη δημοκρατία και δεσμευόμαστε για μια νέα εταιρική σχέση, υποστηρίζοντας ακόμα περισσότερο στο μέλλον τις χώρες εκείνες στην περιοχή, οι οποίες συνεχίζουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ζητήσαμε από την ΕΠΑ το εκπρόσωπο να μεταφέρει το μήνυμα αυτό στην επόμενη επίσκεψη που θα κάνει στην Τινησία και στην Αίγυπτο, τονίζοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαδικασία αλλαγών που λαμβάνει η χώρα. Οι αλλαγές αυτές που έγιναν οδήγησαν σε διάφορες ανακοινώσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το μήνυμα ήταν ένα και το αυτό. Ήταν ότι στηρίζουμε την επιθυμία των λαών για ελευθερία και για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Και αυτό το κεντρικό μήνυμα παγιώθηκε και επανελήφθηκε στην δήλωση που υιοθετήσαμε. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στα άλλα, τα εσωτερικά θέματα που συζητήσαμε. Και πρώτα απ' όλα, και είχε σχεδιαστεί, εδώ και καιρό με δικιά μου πρωτοβουλία συζητήσαμε δύο θέματα τα οποία είναι ζωτική σημασία και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την απόδοση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά τη διαχείριση τη τρέχουσα οικονομική κρίση και να αντιμετωπίσουμε τι μελλοντικέ προκλήσει. Τα θέματα αυτά ήταν η ενέργεια και η καινοτομία. Και τα δύο θέματα αυτά αποτελούν στοιχείο κλειδί για την ευημερία μας. Είναι στοιχείο κλειδί για την Ευρώπη του 2020 και μετά από αυτό. Και για τα δύο αυτά θέματα εμείς θέλουμε να δώσουμε νέα όθηση και υιοθετήσαμε συγκεκριμένες αποφάσεις με συγκεκριμένες προθεσμίες. Προκειμένου να έχουμε μια αγορά της ενέργειας που να λειτουργεί πλήρως, που να λειτουργεί σε δίκτυα και να είναι ολοκληρωμένη θέλουμε να έχουμε μια ενιαία αγορά οι, όλοι είπαν ότι βρισκόμαστε πίσω όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση αν συγκρίνουμε με τον στόχο που είχαμε για 20% για το 2020. Επίσης βρισκόμαστε πίσω και όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη αν συγκρίνουμε με το τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε και πολύ σύντομα με αυτό που γίνεται στην Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια έκθεση πρόοδου όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων που πήραμε τώρα ακριβώ την προηγούμενη εβδομάδα. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να υπογραμμίσω ότι υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Αντιπρόεδρο Σέρκοβιτ, ο οποίο θα πει περισσότερα σε λίγο όσον αφορά την ενέργεια και την καινοτομία. Τέλο, συζητήσαμε την οικονομική κατάσταση. Η ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει να έχει βελτιωθεί πολύ και στην Ευρωζώνη και στις χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετώπισαν πρόσφατα μεγάλες δυσκολίες. Τα σπρέτς έχουν πέσει σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες και οι επιχειρησιακοί δείκτες δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε καλά. Όλοι μαζί πήραμε πρωτοβουλίε πέρυσι και διάφορε ατομικά κυβερνήσει πήραν επίση πρωτοβουλίε και τι εφαρμόζουν. Γνωρίζουμε όμω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν ε, χρειάζεται φυσίχασμό. πήραμε μαθήματα από την κρίση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη στιγμή αυτή για να υιοθετήσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο το Μάρτιο. Και επιτρέψτε μου εδώ να υπογραμμίσω ποια είναι τα κύρια στοιχεία του πακέτου αυτού. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε ισχυρή διακυβέρνηση. Θα έχουμε την έκθεση της Task Force όσον αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς θα το μελατήσετε. Δεύτερον, συγκεκριμένες προτάσεις για να ενισχύσουμε τον μηχανισμό σταθερότητας έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός και να μπορέσουμε να δώσουμε την κατάλληλη στήριξη. Τρίτον, μια τελική απόφαση με δικιά σας γνωμοδότηση όσον αφορά την περιορισμένη τροποποίηση των συνδικών όσον αφορά τον ε, μηχανισμό ε, σταθερότητας. Ελπίζουμε η γνωμοδότησή σας να μας έρθει πριν από το Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου. Τέταρτον, εφαρμογή των προγραμμάτων που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα και την Ιρλανδία. Πέμπτον, εφαρμογή στην Ευρωζώνη μέτρων για να ενισχύσουμε την δημοσιονομική κατάσταση και τέλος για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες να γίνουν δοκιμές αντοχής έτσι ώστε να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση. Για όλα αυτά τα σημεία αποφασίσαμε ποια θα είναι η κατεύθυνση και δώσαμε μια εντολή και κατευθυντήριες γραμμές στους διάφορους φορείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει ολόκληρο το πακέτο στις 24 και 25 Μαρτίου. Οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων των 17 χωρών της Ευρωζώνης συζήτησαν επίσης πόσο να πετύχουμε ισχυρή οικονομική σύγκληση σε συνεργασία μεταξύ μας, ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Αντί να κοιτάμε μόνο το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, του ετήσιου ελλείμματος, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και άλλες πολιτικές που οδήγησαν σε αυτό. Αυτό είναι κάτι νέο. Το ευρώ απαιτεί περισσότερη κοινή πολιτική μεταξύ μας και χαίρομαι που τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι χρειάζεται ισχυρό συντονισμό πέρα από τη μακροοικονομική εποπτεία η οποία αποφασίστηκε με την έκθεση της Task Force. Έτσι ανοίγουν νέοι δρόμοι. Τώρα πρέπει η πολιτική μας βούληση να γίνει πράξη. Σε ποιους τομείς, με τι εργαλεία, με τι περιθώρια και όρια. Και γι' αυτό έδωσα εντολή να υπάρξει διαβούλευση με όλες τις χώρες, με όλους τους γέτες κρατών και κυβερνήσεων, προκειμένου να αποφασίσουμε συγκεκριμένα μέτρα από τώρα μέχρι το Μάρτιο και σε στενή συνεργασία βέβαια με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, μας ενδιαφέρει και η συμμετοχή των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Η έκθεση αυτή θα συζητηθεί μέσα Μαρτίου και από αυτούς. Δεν προτάθηκαν συγκεκριμένε προτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και όπω ε, είπα και στο Λονδίνο πριν από τρει εβδομάδε, ο συντονισμό τη οικονομική πολιτική δεν σημαίνει ομοιομορφία. Τα σημεία κίνηση πολλέ φορέ είναι διαφορετικά μεταξύ του. Πρέπει όμω να πάμε προ την ίδια κατεύθυνση. Είμαι πεπισμένο ότι θα πετύχουμε μεγαλύτερη ακόμα συμφωνία για το πώ θα προχωρήσουμε από τώρα μέχρι το Μάρτιο. Θέλω όμω να υπενθυμίσω σε όλου σα ότι το ευρώ στο σύνολό του εξακολουθεί να είναι ένα ισχυρό νόμισμα. Για 10 χρόνια μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός έμεινε στο χαμηλότερο επίπεδο, μέχρι 2%. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης με τις αποφάσεις που θα πάρουμε το Μάρτιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Αντιπρόεδρος κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. πρώτα του Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ξεκινούμε μέλη του Κοινοβουλίου, καταρχήν θα ήθελα να σα ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Πρόεδρου Μπαρόζο που δεν μπορεί να είναι παρόν στη συζήτηση γιατί είχε ενηλυμένες υποχρέωση μια επίσκεψη με έναν επικεφαλής κράτους αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω κατά τον να σας παρουσιάσω εγώ την θέση της Κομισιόν για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10 Φεβρουαρίου. Όπω συστήσαμε εδώ στο σώμα την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε με πολύ σημαντικά θέματα για το μέλλον τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Οικονομία, Ενέργεια και καινοτομία που ήταν τμήμα τη αρχική υπηρεσία ε, διάταξη, αλλά και η οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά θέματα, γιατί μια οικονομική ανάκαμψη θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση στου πολίτε. Η διάσκεψη κορυφή τη περασμένη Παρασκευή πήρε αποφάσει πολύ συγκεκριμένε με προθεσμίε για δράση για την ενέργεια και την κοινωνία. Οι αποφάσει αυτέ εντάσσονται πολύ καλά στο ευρύτερο πλαίσιο εντατική εργασία για την οικονομική διακυβέρνηση. Ξέρετε ότι η Κομισιόν πρόσφατα δημοσίευσε την πρώτη έκθεση την ετήσια έκθεση για την απασχόληση και ξέρετε ότι προετοιμάζουμε την οικονομική διακυβέρνηση και εργαζόμαστε πάνω στο μηχανισμό οικονομικής σταθερότητας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει την οικονομική διακυβέρνηση και ιδίω στην Ευρωζώνη με θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει αποφασιστικότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων να επιτευχθεί αυτός ο κοινός στόχος. Είναι πάρα πολύ θετικό που τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ε, δεσμεύονται για ευρεία ε, ημερησία διάταξη και ότι πιστεύουν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουν υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Όσον αφορά το νομοθετικό πακέτο, είναι πολύ χρήσιμο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο Εκοφήν να συμφωνήσει πάνω σε μια γενική προσέγγιση με τι αρχέ Μαρτίου. Καλωσορίζει η Κομισιόν επίση τη δέσμευση που ανέλαβε το Συμβούλιο που θέλει να υπάρξει τελική απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί προ τι προτάσει του Κοινοβουλίου που θα βασίζονται στη συνένεση που επετέχθη στην Task Force τη οποία προέδρευε ο πρόεδρο Έρμαν Φαν Η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να βοηθήσει τι συνομιλίε μεταξύ των δύο συνομοθετών μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Εταιρική σχέση, που είναι τόσο σημαντική για την πρόοδο και βέβαια να προωθήσει τον ρόλο της Κομισιόν, καταρχήν πρωτοβουλίας και κατά δεύτερον υποβολή των προτάσεων. Έχει θέσει τα θέματα αυτά για την επόμενη ε, συνεδρίαση του Μαρτίου. Και όσον αφορά και την οικονομική επαγίωση, θέλει η Κομισιόν να τονίσει ότι οι προτεραιότητε αυτέ αφορούν όχι μόνο τα προγράμματα σταθερότητα και σύγκληση, αλλά και τι εθνικέ ε, προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν οι προσπάθειες αυτές να ενταχθούν μέσα στο ευρύ πλαίσιο της στρατηγικής του 2020 που προσπαθούν να προωθούν οι θέσεις απασχόλησης για τους νέους, η παιδεία, η δυνατότητα απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Ευρώπης 2020 είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περαιτέρω βήματα, παραδείγματο χάρη στενότερη οικονομική συνεργασία, θα μπορέσει να ε, βελτιώσει την αγνωστικότητα και την σύγκληση και έτσι να οδηγήσει σε γενικό συνορισμό της οικονομίας. Έτσι ερμηνεύει η Κομισιόν τα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου και θεωρεί ότι συμπληρωματικά βήματα θα πρέπει να εξεταστούν από τις χώρες της Ευρωζώνης για να προωθηθεί η οικονομική συνεργασία και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, πράγμα που θα είναι ευθυγρασμένα με τη συνθήκη. Δηλαδή, θα σεβαστούν τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σεβαστούν την ενιαία αγορά και δεν θα αποκλείσουν τις χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Θα πρέπει να είναι όμως ξεκάθαρο δεν αφαιρούνται αρμοδιότητες από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Κομισιόν χαιρετίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για να ενδυναμώσει την οικονομική συνεργασία για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκριση. Θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη για να είναι σίγουροι ότι όλα αυτά που θα ε, ξεκινήσουν να είναι απόλυτα συμβατά με τη συνθήκη. Όπω είπε ο πρόεδρο Φων Ρόλποη, είμαστε σίγουροι ότι η συνθήκη δίνει επαρκέ πλαίσιο για να προωθήσει την οικονομική ε, διακυβέρνηση. Όπως είπε ο πρόεδρος Φανιλοπόη, θα πρέπει να προχωρήσει σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για να προετοιμάσει η διάσκεψη κορυφή του Μαρτίου. Η Κομισιόν χαιρετίζει τι προσπάθειες που γίνουν να αποχωρήσουν από αυτό που υπάρχει σήμερα επιτάπτω και να βελτιωθούν τα μέτρα για την πρόθεση τη ευρωπαϊκή αναγνωστικότητα. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και να γίνει ταυτόχρονα σεβαστός βέβαια ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έρχομαι τώρα στην ενέργεια και στην καινοτομία. Κεντρικό μα στόχο είναι η αποκατάσταση τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητά μα. Α μην ξεχνάμε ότι η ενέργεια και η καινοτομία είναι επίση δύο τομεί όπου η κοινοτική προσέγγιση και η ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να προσφέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Το πρώτο ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ενέργεια έθεσε συγκεκριμένου ε, στόχους και επιδόσεις. Χρειάζεται να επιταχύνουμε για να φτάσουμε στους στόχους μας για το κλίμα και για την ενέργεια, ε, ε, επάρκεια, έρευνα και ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι συμπληρώνονται από την εξωτερική διάσταση τη ενεργειακής πολιτική, όπου τα κράτη-μέλη έχουν τώρα συμφωνήσει να μοιράζονται τι πληροφορίε όσον αφορά τι εξωτερικέ συμφωνίε για την ενέργεια. Όπω υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα, ότι η αύξηση τη επάρκεια στην ενέργεια σημαίνει περιορισμός της ε, κατανάλωσης ε, για τις ε, βιομηχανίες και για τους ιδιώτες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε σαφές μήνυμα για την αύξηση της ενεργειακής επάρκειας, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. Πλήρως ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά είναι απαραίτητο προϋπόθεση για την αλληλεγγύη και την ασφάλεια στην, στον ανεφοδιασμό. Επίσης, σημαντικό μήνυμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το 2014 μέσω της άρσης όλων των τεχνικών και των ρυθμιστικών φραγμών. Αυτό θα αποδεσμεύσει τεράστιο δυναμικό για την ανάπτυξη και αν τα καταφέρουμε σωστά οι καταναλωτέ θα εξοικονομήσουν 30 δις ευρώ ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ηλεκτρισμό από πιο φθηνές πηγές. Υποδομές και εντοπισμός κατάλληλων μέσων χρηματοδότησης στα τα κράτη-μέλη να μην απομονώνονται από την ευρωπαϊκή αγορά. Μέχρι το 2015 η Κομισιόν θα καταθέσει σχετικές προτάσεις φέτος για την διευκόλυνση των επενδύσεων σε υποδομές. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στις, στις ασφαλείς, ε, ε, στον ασφαλή άνθρακα η δέσμευση για ενθάρρυνση της εξωτερικής πολιτικής ε, σε σχέση με την ενέργεια είναι ακόμα ένα αποτέλεσμα, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμείς θα παρουσιάσουμε ε, ανακοινωθέν για την εξωτερική πολιτική ενέργειας ε, αργότερα μέσα στο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει την ε, καινοτομία ΔΕ στην αιτήσια της έκθεση για την ανάπτυξη, ε, στο επίκεντρο μάλλον της έκθεσης αυτής. Η πρόκληση είναι τώρα να προχωρήσουμε στην φάση ε, των επιδόσεων, εντοπίζοντα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αυτό ακριβώς κάνουν και αυτό το καλωσορίζουμε η Κομισιόν κάλεσε το Συμβούλιο να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική όσον αφορά την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μα ακολούθησε εδώ και επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλε προποθέσει ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για του επενδυτέ στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτό σημαίνει καθεστώ πνευματικών δικαιωμάτων πιο αποτελεσματικό, καθεστώ κρατικών προμηθειών που θα προωθεί την καινοτομία και πιο γενικά απλοποίηση των κανόνων και τη κατάργηση της γραφειοκρατίας. Μια προεγνήσια δε ευρωπαϊκή αγορά για τα επισφαλή κεφάλαια και για το ψηφιακό περιεχόμενο. Όλα αυτά τα υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ε, ταχύτατα θα ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος για την Αίγυπτο να πω μετά από τα όσα πολύ ωραία μας εξέθεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα της Αιγύπτου και της Τινησίας αύριο συλλογικά στην Κομισιόν και αν θέλετε κάτι να προσθέσω στο τέλος. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρος, ο κύριος Ζωζεφ Ντόλ από το ΕΛΚ τώρα έχει το λόγο εκ των πολιτικών ομάδων. Αρχίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φανερομπάου, κύριε Αντιπρόεδρε Σέρκοβιτς, μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρησιμοποίησατε τρεις λέξεις κλειδί. Φιλοσοφία για την ενέργεια, ανησυχία για την Αίγυπτο και αποφασιστικότητα για τη διακυβέρνηση. Θέλω να επανέλθω σε αυτά τα τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα για την ενέργεια. Οι 27 δήλωσαν ότι καμία χώρα μέλος δεν πρέπει να μείνει απ' έξω μέχρι το 2015 όσον αφορά το ενεργειακό επειδή δεν έχει τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Συμφωνώ με τη φιλοδοξία αυτή και χαίρομαι που ελήφθησαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν γιατί τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να απομονωθούν για ένα τόσο στρατηγικής και μεγάλη σημασία θέμα αλλά ούτε πρέπει να εξαρτώμαστε απ' έξω για την ε, ενεργειακή μας προμήθεια. Η λύση δεν είναι λιγότερη Ευρώπη, είναι περισσότερη Ευρώπη. Το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Την Παρασκευή οι επικεφαλείς κρατόκια και κυβερνήσεων συμφώνησαν ε, λοιπόν ε, για την αγορά ενέργειας. Είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν, μια που είναι τα ίδια τα κράτη-μέλη που έχουν θέσει τους κανόνες. Και έτσι είναι απόλυτα φυσιολογικό τους κανόνες αυτούς να τους κάνουν πράξη και για την ενέργεια αλλά και για το σύμφωνο σταθερότητας όπου οι κανόνες πρέπει να μπαίνουν σε εφαρμογή. Και αν δεν μπαίνουν σε εφαρμογή τότε η Επιτροπή, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, είμαι εδώ για να σας το υπενθυμίσω και εσείς πρέπει να το υπενθυμίζετε στα κράτη-μέλη, εφόσον χρειάζεται, αν δεν τηρούν τους κανόνες, τότε πρέπει να τους πάτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας τώρα. Συγχαίρω το Συμβούλιο που έκανε ένα βήμα προς τα μπρος προωθώντας τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και στις τεχνολογίες της ασφαλής με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Όντω πρέπει σε αυτέ τι ενέργειε να βασιζόμαστε. Καιρό ήταν να έχει το πολιτικό θάρρο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να το πει. Όσον αφορά τώρα την Αίγυπτο και την κατάσταση στην Μεσόγειο, στου εταίρου μα. Και με ανησυχεί η κατάσταση. Ίσως όμως όχι μόνο για τους ίδιους λόγους που υπενθύμησε ο πρόεδρος Φανροπάου, γιατί εμένα το πρώτο που με ανησυχεί είναι το ότι η Ευρώπη, που είναι ο πρώτος δωρητής, δεν καταφέρει να μιλήσει με μία μόνο φωνή. Για άλλη μια φορά. Έχουμε μία είπατε εκπρόσωπο, όμως τα κράτη-μέλη είναι τελικά εκείνα τα οποία ε, βγάζουν ανακοινοθέντα προς πάσα κατεύθυνση και με διαφορετικό τρόπο για τις εξωτερικές υποθέσεις. Για τους Ευρωπαίους δεν πρέπει να φροντίσουμε να μας σέβονται περισσότερο, οι εταίροι μας να μας ακούνε περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα γίνει. Και εγώ και η ομάδα μου το ίδιο πιστεύει. Γιατί για άλλη μια φορά η λύση δεν είναι λιγότερη Ευρώπη, αλλά περισσότερη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να μιλάει ενωμένη, με δυνατή φωνή, που φροντίζει να ακουστεί το μήνυμά τη, να ακουστούν οι αξίε τη και ευαισθησίε τη. Αυτό θα έπρεπε να ήταν και ένα από τα επιτεύγματα της Λισαβόνα. Επούντο. Έτσι λοιπόν, Πρόεδρε, ρωτάω και ρωτάω και εσά, κύριε Πρόεδρε, πού είναι. Τέλο, για την οικονομική διακυβέρνηση. Επ' αυτού, κύριε Πρόεδρε, Εκφράσατε την ικανοποίησή σας για την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εγώ θα βάλω εδώ μια μικρή απόχρωση, διότι χαίρομαι μεν που το θέμα της διακυβέρνησης και της δημοσιονομικής σύγκλησης, αλλά και της φορολογικής και της κοινωνικής δεν αποτελούν πια ταμπού, αλλά συγχρόνως πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστούν, να συζητηθούν σε ένα πλαίσιο που να μην είναι καθαρά εθνικό, διακυβερνητικό, αλλά κοινοτικό. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, σωστό είναι στις ευρωπαϊκές συζητήσεις να μπαίνουν θέματα τόσο σημαντικά όπω είναι η ηλικία ε, η διάρκεια εργασία, η αναπροσαρμογή των μισθών ή το δημόσιο χρέο και να μπαίνουν στα συντάγματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Εξάλλου, είναι θύματα είναι θέματα συγγνώμη, για τα οποία οι πολίτε μα συζητούν εδώ και καιρό. Για όλα όμω αυτά τα θέματα πρέπει να συζητάμε και να αποφασίζουμε χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι επιβάλλουμε, αλλά ότι βάσει της κοινοτική μεθόδου συζητούνται και αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέθοδος αυτή έχει αποδείξει την αξία της. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω ότι η λύση δεν είναι περισσότερη αντιπαράθεση μεταξύ των χωρών μελών, όχι περισσότερες κοινέ αποφάσεις. Πρέπει να συζητάμε για τα πράγματα που μας ενοχλούν, κοινωνικές, ρυθμίσεις, φορολογικές κτλ. Γιατί χωρίς αυτά δεν θα υπάρχει αλληλεγγύη που να τη δέχονται οι πολίτες μας και να φροντίζουν να υπάρχει. Και χωρίς αλληλεγγύη δεν θα υπάρχει Ευρώπη. Οι χώρες μας πρέπει να είναι αποφασισμένες να τηρήσουν τους κανόνες διακυβέρνησης, διότι χρειάζονται, μας το απέδειξε αυτό η κρίση, και είναι και απόλυτη αναγκαιότητα όμως η αποφασιστικότητα πρέπει να είναι εξίσου μεγάλη για να τηρούνται μαζί επίσης ώρες για όλους και με αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. E, Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κ. Μάρτιν Σούτς έχει το λόγο. Εξονόματος της σας ομάδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Κοιτάξτε, μου δώσανε εδώ πέρα από το λάθος ταβέρνα. Δεν είμαι ο Βέσουρτ εγώ, δεν ξέρω ποιο είναι Βέ, Βλαδίμηρο, ξέρω εγώ πώ τον λένε. Εγώ δεν είμαι αυτό πάντω. Εμένα με λένε Μάρτιν, Μάρτιν Σούλτ. Uh, Πρόεδρε, δεν μπορώ να είμαι τόσο το προς εσάς όπως ο, ο, ο Ζωζεφ Βόλ παρόλο που ήταν πολύ τολμηρή η ομιλία του γιατί αν τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με ευρεία πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει πάνω σε κάποια σημεία που συζητήσαμε, ακόμα καλύτερα. Κύριε Ρομπάη, μετά από το Συμβούλιο αυτό αναρωτιέμαι πραγματικά ποιο είναι το δικό σας έργο. Εσάς το έργο σας είναι να κρατήστε ενωμένο το Συμβούλιο και να το εκπροσωπείτε στο σύνολό του. Εγώ έτσι κατανόησα τουλάχιστον τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αλλά βλέπω όμω ότι η κυρία Μέρκελ και ο κύριο Σαρκοζή έχουν τελείω διαφορετική άποψη. Τι έγινε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρχίσω και εγώ με την Αίγυπτο, όπω και εσεί κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. γιατί αυτό που κάνουμε είναι να μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Στη Mappen Show υπάρχει μια, μια εικόνα όπου είναι δύο ηλικιωμένοι κύριοι που κάθονται στο μπαλκόνι, σχολιάζουν τα πάντα αλλά δεν τους λαμβάνει κανένα σοβαρά υπόψη του. Αυτό περίπου είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική. Το είπα ήδη την περασμένη εβδομάδα εδώ. Εκφράζεστε εσεί, ο κύριος Μπαρόζο εκφράζει την άποψή του, ο κύριος Σαντών, μετά ξεχωριστά ο κύριος Σαρκοζή, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Κάμερον και άλλοι ίσως και εμείς. Δεν ωφελείστε τίποτα όμω. Νομίζω ότι η στάση της, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι πιο δυσνόητη από ότι αυτά που γίνονται στην Αίγυπτο εάν δεν καταλάβουμε κύριε Πρόεδρε ότι αυτά που γίνονται εκεί είναι δική μας πολιτική δεν θα προχωρήσουμε. Γείτονα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όχι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Έχουμε ιστορικού δεσμού προ την Αίγυπτο που δεν εκμεταλλευόμαστε. Και έχουμε και ένα συμφέρον ασφαλεία που δεν εκφράζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δράσει εδώ. Πάρα πολύ λυπηρό μου φαίνεται. Και σας το λέω εγώ, το είπα και στην Καθιέστον Θα περίμενα να έχει πάει εκεί. Να μιλήσει εκεί επί τόπου με τις δυνάμεις που δημιουργούν. Γιατί είναι μια πραγματική μοναδική ευκαιρία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που είναι εκεί κάτω οι άνθρωποι δεν θέλουν θεϊκό κράτος, ίσως δεν θέλουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορούμε όμως να τους παρουσιάσουμε τις αξίες της Ευρώπης, να τους στηρίξουμε, να ε, ε, ακολουθήσουν. Αυτό θα ήταν ίσως το πρωταρχικό μας έργο. Γιατί το συζητάει αυτό το Συμβούλιο ή αν το συζήτησε γιατί δεν μας το λέει. Μετά, όσον αφορά το σύμφωνο για την αναγωνιστικότητα που τα συζητήσαμε, Έχω να σας πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι συμφωνία για αναγνωστικότητα. Είναι μια προσπαθία της Ομοσπονδικής Δημοκρατία της Γερμανίας να επιβάλλει ένα πρόγραμμα λιτότητα στην Ευρώπη. Και θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Πιστεύει πραγματικά κανένα σοβαρά ότι μπορούμε, αν καταργήσουμε το, το σύστημα αυτό με τις προσωπικές των μισθών σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιέσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι σφαλμένο γιατί θα υπάρχουν στρεβλώσεις κοινωνικές. Στι πολλέ χώρε που έχουν διαφορετικό σύστημα από τη στη Γερμανία, η αυτόματη τιμορυθμική προσαρμογή είναι η μόνη δυνατότητα να εγγυηθούν μια σταθερότητα εισοδήματο για του πιο αδύναμου. Άμα γίνει αυτό, εσεί ήσασταν πρωθυπουργό μια χώρα που ακριβώ αυτό κάνει. Ε, θαυμάσια άμα πάνε έτσι τα πράγματα. Θα έχετε άλλη μια κρίση, χωρά τη άλλη που έχετε ήδη στη χώρα σας. Μετά, ελάχιστο ποσοστό για επενδύσεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στην παιδεία και στις υποδομές εκατό του ΑΕΠ. Η... Αυτό αναφέρεται στο σύμφωνο ανταγωνισμού. Πολύ καλό μου φαίνεται αυτό. Έρευνα, ανάπτυξη, παιδεία και υποδομή. Αυτό εκεί χρειάζονται επενδύσεις που θα προωθήσουν την ανάπτυξη. Οι ίδιοι όμω που αποφασίζουν αυτά, κύριε Σέκβος, κύριε Φανρόποη, είναι εκείνοι που στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να κάνουν περικοπέ ακριβώ αυτού τους τομείς. Και α με εξηγήσει κανένα πώς μπορούμε έτσι να προωθήσουμε την Ευρώπη. Δεν είναι ασφαλμένη η άγουσα αυτή είναι πρόγραμμα λιτότητας. Δεν είναι πρόγραμμα ε, βα, ε, ανάπτυξης αηφόρου. Και τέλος, είναι ένα πρόγραμμα που διαχωρίζει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει με τους 27 ή θα αποτύχει. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο για μας. Γι' αυτό είμαι, είμαι ευγνώμων προς τον Ιώζεφ Τόλ. Γιατί εάν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε αυτό, αυτό το κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα τοποθετεί έτσι όπως το έκανε υπάρχει ένα, ένα όργανο στο οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίφερ Χόφσατ, πρόεδρο των Φιλευθέρων, παρακαλώ. Uh, yes, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ασχοληθώ μόνο με το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και θα ξεκινήσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Σούλτς. Και αυτή είναι η πρώτη μου ανησυχία. Έχω τρεις, αλλά αυτή είναι η πρώτη. Ότι στο δεύτερο πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση που βρίσκεται σήμερα τάπητος μετά την ε, διάσκεψη είναι πάλι με την διακυβερνητική μέθοδο. Αυτή χρησιμοποιείται. Και το γαλλογερμανικό σύμφωνο. Αυτή η διακυβερνητική μέθοδος, το ξαναλέω, δεν λειτουργήσε στο παρελθόν ούτε θα λειτουργήσει και στο μέλλον. Δεν λειτουργήσε στο παρελθόν, συνάδελφοι. Για τη σταθερότητα και ανάπτυξη, για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Γιατί ούτε η Γαλλία και η Γερμανία δεν το κατάφεραν. Ούτε με την Λισαβόνα, με τη στρατηγική της Λισαβόνας δούλεψε η διακυβερνητική μέθοδος. Όχι. Και τότε χρησιμοποιήθηκε η διακυβερνητική στρατηγική και δεν λειτουργήσε κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι η ανησυχία μου, ότι αυτή είναι και η αδυναμία του πακέτου που συζητιέται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χθε ο κύριο Τρισέ ήταν στη διάσκεψη των Προέδρων, το είπε και ο κύριο Βέμπελ. Συνήθω ο κύριο Βέμπελ και ο κύριο Τρισέ δεν λένε τα ίδια, αλλά για αυτό το θέμα είπανε το ίδιο. Είπε ότι οι ελλείψεις της μεταρρύθμισης που βρίσκεται μπροστά μας σήμερα είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο από το Συμβούλιο και αυτό δεν δουλεύει. Και ένα άλλο παράδειγμα, συνάδελφοι. Μπορείτε να φανταστείτε ότι οι κανόνε ανταγωνισμού στην Ευρώπη θα έπρεπε να ήταν αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μπορείτε να φανταστείτε κάτι τέτοιο, να είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μα τότε ποτέ καμία κυβέρνηση δεν θα έχει δεχτεί τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε και να επαναλάβουμε. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν πιστεύουμε στην διακυβερνητική προσέγγιση που αποτελεί και τη βάση του λεγόμενου γαλλογερμανικού συμφώνου. Η δεύτερη τώρα ανησυχία μου έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη, συνάδελφοι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία, μυστική συμφωνία που λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία για να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Αυτό Μείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία για το γαλλογερμανικό πακέτο, ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο μεταξύ του. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εδώ πέρα παίζουμε με τη φωτιά. Η τρίτη μου ανησυχία είναι, Πρόεδρε, ο τρόπος με τον οποίο έχει προχωρήσει αυτή η γαλλογερμανική πρόταση, πώς προτάθηκε. Για μένα είναι καταστροφή αυτό. Πήρα το κείμενο. Να, όταν κάποιος ε, συνεργάζεται με την GDU στη Γερμανία, το παίρνει. Λοιπόν, σε 24 ώρες, εσείς δεν το πήρατε, ε, δεν το πήρες, λυπάμαι. Εγώ όμως το πήρα πριν ξεκινήσει το Συμβούλιο, 24 ώρες πριν ξεκινήσει το Συμβούλιο, στα γερμανικά, να το. Και σας λέω ότι πολλοί συνάδελφοι στο Συμβούλιο και οι Γερμανοί ξεκίνησαν το Συμβούλιο χωρίς να έχουν στα χέρια τους το κείμενο αυτό, έτσι όπως προτάθηκε. Και εδώ το λέω, δεν είναι δυνατόν στο μέλλον η οικονομική διακυβέρνηση εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη και η πρόταση να έρχεται από την Κομισιόν και από πουθενά άλλου. Και, τελειώνω με αυτό πρόεδρε, είδα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τελικά κάνει έναν διεθνή οργανισμό Ευρωπαϊκών Εθνών την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο. Κακός. Δεν είναι έτσι που πρέπει να προχωρούν τα κοινοτικά θέματα. Κύριε president συμπρόεδρος των Πρεσίνων. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριοι πρόεδροι, οι συνάδελφοι ήδη εξέφρασαν την ατμόσφαιρα που υπάρχει στους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων μετά τη διάσκεψη κορυφής. Πολύ καλά την παρουσίασαν και θέλω να τονίσω ένα πράγμα μόνο. Σιγά σιγά για μένα είναι ανησυχητικό ότι μετά από δια... κάθε διάσκεψη ε, κορυφής άσχετα πόσο πτωχά είναι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται δημοσίως μετά από κάθε διάσκεψη κορυφής παίρνουμε εκθέσεις σαν όλα να ήταν θαυμάσια και καταπληκτικά. Αυτό μου θυμίζει ανακοινωθέντα από ε, κεντρικά, κεντρικά γραφεία κυβερνήσεων όταν τα πράγματα δεν ήταν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώς πραγματικά καταλούν λίγο στο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Μάρτιν Σούλτς. Πολιτικά συστήματα που δεν συζητούν ειλικρινά τα προβλήματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Για τα επιμέρους προβλήματα τώρα έχω να πω Αίγυπτος. Ντροπή. Μια μέρα ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση η διάσκεψη κορυφής αυτή. Αισθάνονται οι άνθρωποι εκεί ότι τους έχει εγκαταλείψει η Ευρώπη. Θεωρούν ότι πραγματικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει νέα κυβέρνηση στην Αίγυπτο με αυτόν τον δικτάτορο που έχει οριστεί από τη Δύση εκεί και θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενέργεια. Επρόκειτο για διάσκεψη κορυφή ενέργεια. Θα πρέπει ε, ακόμα και σήμερα να ζητήσουμε συγγνώμη πως το αποκαλούσαμε διάσκεψη κορυφή ενέργεια. Γιατί προχωρήσαμε ίσω κάποια χιλιοστά όσον αφορά τι απαραίτητε βελτιώσει τη υποδομής. Πραγματικά όμως αποτελέσματα δεν ε, μας έφερε αυτή η διάσκεψη κορυφής. Το είπα ήδη και στο Στρασβούργο ότι νομίζω ότι με τον Επίτροπο Πίμπαλξ είχαμε προχωρήσει ε, έτη φωτός και ότι το περασμένο έτος της Βρυξέλλης ήταν απώλεια. Όσον αφορά το γερμανογαλλικό σύμφωνο, έχω την εντύπωση αυτός ο τίτλος που χρησιμοποιείται τώρα, αντί αυτού που συζητείτε, δηλαδή εμείς συζητάχαμε κανονικά για ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση. Και αυτός ο τίτλος πραγματικά που δεικνύει όλη την καταστροφή που έφεραν η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή. Και δεν καταλαβαίνω γιατί καμία κριτική η οποία ε, παρουσιάστηκε από του αρχηγού των κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της ε, διάσκεψη κορυφή, καμιά από τι επικρίσει αυτές δεν παρουσιάστηκε ούτε από εσάς, κύριε Φανερόμποη, ούτε από την Κομισιόν. Κρυφτούλη παίζεται. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν θα μα βοηθήσει να φτάσουμε σε καλό αποτέλεσμα. Και θα ήθελα τελειώνω να σας πω ότι τελικά δεν πιστεύω ότι η κοινοτική μέθοδος κατανοείται στο Συμβούλιο και αυτό είναι λιγάκι και απολογισμό της δικής σας εργασίας κύριε Φανελόπολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τίμωθη Κύρκοβ έχει το λόγο. Uh, Πρόεδρε, η ελευθερία είναι μια αξία την οποία, η οποία είναι κοινή για όλου εδώ και για τη δική μου ομάδα είναι από μια από τις πιο σημαντικές αρχές. Πιστεύουμε ότι η μεγιστοποίηση της ατομικής ελευθερίας στην κοινωνία περιορισμένο κράτος και χαμηλή φόρη είναι ο καλύτερος τρόπος για τους, την επίτευξη των κοινωνικών, των, των οικονομικών και των πολιτικών ε, στόχων. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε τις εξελίξεις στην Ισία, την οποία επισκέφτεται ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, στην Αιγύπτο και ως ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, πράγμα το οποίο υποστηρίζουν και τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της τελευταίας ε, Παρασκευής. Είναι μύθος για όσους θέλουν να ελέγχουν την πολιτική, τους πολίτες τους, ότι η δημοκρατία είναι ασύμβατη με το Ισλαμικό κράτος, με την αραβική κοπολιτισμό. Τι πρόσφατε εξελίξει έδειξαν πω και οι αραβικοί λαοί έχουν την ίδια επιθυμία για ελευθερία και δημοκρατία. Η καταπίεση έχει πνίξει την οικονομική ανάπτυξη και οι λαοί τη Βορείου και τη Μέση Ανατολή έχουν ε, υποστεί καταστολή και έχουν μείνει πίσω. Η οικονομική του ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανεργία και από μεγάλε κοινωνικέ αναταροχέ, ε, Πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει στη γέννηση κάποιων ακραίων ομάδων. Όμως ε, ε, η μεγάλη πλειοψηφία δεν θα ακολουθήσει αυτό το ε, δρόμο. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την διαδικασία μετάβαση στην Αίγυπτο. Θα πρέπει ωστόσο να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Μουμπάρακ ήταν ένα μεγάλο Αιγυπτιος πατριώτη, φίλος της Ευρώπης και της Αμερικής, επιδίωξε την ειρήνη με το Ισραήλ και σίγουρα γι' αυτό έχει σώσει ζωέ. Δεν μπορούμε ωστόσο να είμαστε τυφλοί στην, αυτο, στην αυταρχική φύση του καθεστώτο του και πλέον είναι η ώρα για την αλλαγή. Αυτό θα πρέπει να γίνει μετάξυ. Ξέρουμε μετά από την εμπειρία μα εδώ στην Ευρώπη πως η δημοκρατία έχει κάθε ευκαιρία για επιτυχία αν βασιστεί σε ένα λειτουργικό κράτος το οποίο μεταμορφώνεται με βασι... με σταδιακά για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των λαών. Και ξέρουμε από την επανάσταση του Ιράν ότι μια σύντομη στιγμή ελευθερίας μπορεί πολύ βία να πνιγεί από ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο αρπάζει την εξουσία από ένα άλλο αυταρχικό καθεστώς. Άρα λοιπόν για την ε, Αίγυπτο και την Μέση Ανατολή και για τη Λευκορωσία τις οποίες οι πολίτες ε, τώρα τραγικά είδαν να τους αρνούνται το δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σταδιακά. Καλωσορίζουμε το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την επιδίωξη της οικονομικής ελευθερίας και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για την καινοτομία. Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς για την έρευνα και την καινοτομία χρειάζεται υποστήριξη όπως και η ενιαία αγορά, η ψηφιακή, καθώς και η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ενεργειακής αγοράς για να προωθηθεί η επάρκεια σε ενέργεια. Όμως προσοχή, είναι σωστό να καταργούνται τα τεχνητά εμπόδια στο εμπόριο και την κοινοτομία. Θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να παρέμβουμε στην αγορά για, κανονισμού. κανονισμούς. Ε, σε αυτό το τομέα, Πρόεδρο, όπω και στου άλλου οι κυβερνήσει θα πρέπει να θεσπίσουν τα κατάλληλα νομικά και πολιτικά πλαίσια, να δώσουν το κατάλληλο κλίμα και κίνητρα για επενδύσει, και έπειτα να επιτρέψουν στι επιχειρήσει, του επενδυτέ του εφευρέτες και τι επιχειρήσει να επεκταθούν. οικονομική ελευθερία και όχι και παρέμβαση θα ανοίξει το δρόμο για όλη την μελλοντική μας ευημερία. Σας ευχαριστώ. κυρία Μαρίζα Ματίας από την ε, Ενωμένη Ιστερά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, εκφράζοντας μάλλον την ε, λύπη μου ε, σε σχέση με τα όσα ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, γιατί σε αυτό το Συμβούλιο που έπρεπε να είναι ευκαιρία όπου θα έπρεπε να συζητηθούν τα θέματα για την ενέργεια, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης ε, κατέληξε να συζητά μόνο για την ασφάλεια και για τέτοια θέματα. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για την ενέργεια ως ε, τρόπο για δημιουργία θέσης απασχόλησης Έχουμε γκρίνει ένα σωρό σχετικά έγγραφα και όσον αφορά και μόνο και μόνο αν μιλούσαμε για την επάρκεια την ενεργειακή των κτηρίων θα μπορούσαμε άμεσα να ενεργήσουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Έγινε μόνο μία ε, δήλωση ενδιαφέροντος. Ωστόσο θα πρέπει να μπορέσουμε να λύσουμε ικανοποιητικά τα προβλήματα τόσο με βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι η ανανέωση του οικονομικού κόσμου, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και δεν ε, φτάνει να το σκεφτόμαστε μόνο για το μέλλον, πρέπει να το σκεφτούμε και για σήμερα. Ε, και σκέφτομαι αυτές τις ευρωπαϊκές ε, χώρες που αφισβητούν την γερμανική πρόταση όσον αφορά τους μισθούς και τον πληθωρισμό γιατί οι χώρες οι πιο περιφερειακές αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την μείωση των μισθών. Αυτή η γαλλογερμανική πρόταση ή όπως η γερμανική πρόταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια οικονομική πρόταση που στην ουσία εμβαθύνει και αυξάνει την ε, απόκληση ανάμεσα στις χώρες του κέντρου και της ε, περιφέρειας και δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα. Καταρχήν γιατί χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να μειωθεί το χρέος. Μπορεί να ε, μειωθεί το έλλειμμα, αλλά όχι το χρέος. Και το έλλειμμα είναι το βασικό πρόβλημα της οικονομίας των περιφερειακών χωρών. Αυτό θα έπρεπε να υπάρξει, γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική, μόνο και μόνο για αυτό το θέμα. Αυτό το μοντέλο είναι λάθος η Γερμανία δεν μπορεί ε, να είναι μόνο ε, εκείνη που προτείνει συγκεκριμένα μοντέλα επιβάλλοντας κυρώσεις σε όλους τους άλλους θεωρώ πως κάτι είναι πάρα πολύ άδικη θα πρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ουσιαστική να μην επικυρώνει μόνο τις συλλημμένες αποφάσεις της Washington αυτό σε, θέμα, σε σχέση με την Αίγυπτο ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φάρατζ, Ελευθερία και Δημοκρατία Κύριε Φανόπη εκεί που μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι ε, συνθήκες επικροτούν στην ε, ζωή της Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα, η κοινή γνώση είναι, γνώμη είναι αυτό. Καμιά φορά μάλιστα οι ε, εκλογές καταψηφίζουν συνθήκες. Παρ' όλα αυτά το ξεπεράσει τα προβλήματα. Η κυρία Μέρκελ βέβαια είχε ένα πραγματικό πρόβλημα. Χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 122 για τα καμβόλια για την Ιρλανδία και την Ελλάδα και είναι σαφές ε, ότι αυτό ήταν παράνομο. Το ξέρουμε όλοι, δεν τον επέτρεπαν οι συνθήκε. Λοιπόν, οι τέσσερις ε, ε, καθηγητές της, Γερμανίας που την προ, ναι, στα δικαστήρια την έκαναν να ζητάει τώρα να αλλάξει συνθήκη. Χρειαζόμαστε, λέει, τώρα ένα μόνιμο ε, μηχανισμό σταθερότητα. Αυτό δεν με κάνει να εμπνέομαι από εμπιστοσύνη, γιατί αυτό νομίζω καθυστερεί τον κατακαιρματισμό τη Ευρώπη. Παρ' όλα αυτό, αποφασίστηκε να αλλάξει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Υπήρξε όμω και μια άλλη πρόκληση για τη συνθήκη. Δεν το ακούσατε ίσω ακόμα, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο τις πέντε εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση για μια απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει οι φυλακισμένοι να ψηφίζουν. Ε, δεν, ίσως δεν το πιστεύετε, αλλά οι περισσότεροι ε, Βρετανοί εκλογεί δεν συμφωνούν. Ακόμα μάλιστα, ακόμα μάλιστα και οι βουλευτές αισθάνονται έτσι και την Πέμπτη το βράδυ θα υπάρχει ελεύθερη ψηφοφορία στο Westminster και φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία ε, Βρετανών βουλευτών θα καταψηφίσουν την ιδέα να έχουν δικαίωμα ψήφου οι ε, φυλακισμένοι. Και αυτό θα ήταν η πρώτη πρόκληση του, Ευρωπα... του Βρετανικού, της Βρετανικής Βουλής στη Συνθήκη της Αβώνας. Γιατί λέει ο, το, συνθή, το άρθρο 6 ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία και που θα μπορούσε δηλαδή ο κύριος Κάμερο να έρθει την επόμενη φορά να ζητήσει όπως η κυρία Μέρκελ να αλλάξει συνθήκη. Δεν ξέρω αν θα έχει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας θα ξανανοίξει τώρα στην Βρετανία και θα πρέπει να γίνει μια, ένα δημοψήφισμα και θα ήταν καλό νομίζω να σας πω αυτά τα καλά νέα σήμερα. Έτσι φαντάστηκα. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φίλιπ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Με αναμειγμένα συναισθήματα κοιτάει ο κόσμος τα όσα έγιναν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και τα όσα διεξήχθησαν στο περιθώριο του Συμβουλίου αυτού. Ορισμένες χώρες, οι μεγάλες, μεταξύ τους, από ό,τι φαίνεται, προσπαθούν να αποφασίσουν ποια μέτρα θα πρέπει να αναλάβουν οι υπόλοιπε χώρες μέλη. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Ακούσαμε εδώ για τη μέθοδο. Κατά πόσο είναι η κοινοτική, η διακυβερνητική μέθοδος η οποία είναι κατάλληλη για να λυθούν τέτοια προβλήματα που έχουμε στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να είναι η Γαλλία και η Γερμανία που να τα αποφασίσουν. Περισσότερη σύγκληση είπαμε ότι χρειάζεται, περισσότερη συμμετοχή των πολιτών και περισσότερη φορολογική πολιτική και πολιτική μισθών. Τι πάει στραβά στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να δούμε τι γίνεται στις πιο δύναμε οικονομικά χώρες. Πρέπει να βασιστούμε στη δικιά τους κατάσταση και στις δικές τους ανάγκες. Είναι δυνατόν να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών όσον αφορά τη φορολογική πολιτική και την πολιτική μισθών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πάντα ότι ο ανταγωνισμός χρειάζεται για την ευημερία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το λαμβάνουμε αυτό πια υπόψη μας. Είμαστε σε κρίση και συνήθως όταν είμαστε σε κρίση αφήνουμε στην πάντα όλα τα άλλα προβλήματα εναρμόνιση των φορολογικών ε, πολιτικών μιλάμε. Μιλάμε για, τους, ε, για τον ευρωπαϊκό φόρο και γενικά για διάφορες λύσεις θαύμα που προσπαθούμε να βρούμε. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία και αυτό σημαίνει περισσότερη κεντρική κατεύθυνση όλων. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα επικεντρωθώ και θα είμαι σύντομος. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στα δύο θέματα τα οποία ακούσαμε πολύ εδώ σήμερα και θα αφήσω στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να απαντήσει για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και την καινοτομία. Λοιπόν, για τη συζήτηση σχετικά με τόσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο και όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε από δύο οπτικές γωνίες. Απ' τη μια είναι το θέμα του περιεχομένου και απ' την άλλη έχουμε την οπτική γωνία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και της διαδικασίας. Τόσα άκουσα σήμερα είχαν να κάνουν περισσότερο με το δεύτερο θέμα. Και λυπούμε γι' αυτό, ειλικρινά διότι θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, ακόμα και αν είναι σύντομη, επί του περιεχομένου. Δηλαδή τι προτάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε την ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά την Αίγυπτο και την οικονομική διακυβέρνηση. Όμως άκουσα περισσότερο να μιλάτε για τη διαδικασία. Λοιπόν, για την Αίγυπτο ας ξεκινήσω. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Δεν ξέρω τι συνέβαινε πάντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όταν ακούω αυτά που λέγονται στην Ευρώπη μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η Αίγυπτος ήταν πλήρως απούσα. Δεν ακούγαμε τίποτα για την Αίγυπτο σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα. Μιλάω γενικά τώρα, έτσι, γενικά. Προτιμούσαμε τη σταθερότητα, μια σταθερότητα η οποία βέβαια απέφερε καρπούς και ορισμένοι από εσά είπαν πόσο πολύ έχει συνεισφέρει η Αίγυπτος στη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Όμως η σταθερότητα έκρυβε ακινησία και έλλειψη αηφορίας. Διότι δεν μπορεί να παραβιάζουμε την ε, κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία για πάντα. Και έτσι ο Αιγυπτιακός λαός μίλησε δεν περίμενε τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου και δεν θα τις περιμένει. Ούτε την Ευρώπη, ούτε τις Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε κανέναν άλλον. Οι οποίοι βρέθηκαν εξαπρόπτου με αυτά που έγιναν, γίνονται και θα γίνονται στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν είναι οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι που μιλάνε. Και είναι οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι κατά κάποιο τρόπο που θα αποφασίσουν για την τύχη τους. Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε από την Ευρώπη με θετικά μηνύματα. Και το κάναμε αυτό. Βέβαια, από διάφορες πλευρές χωριστά. Συμφωνώ. Όμως, αν τα βάλουμε δίπλα όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία δημοσιεύτηκαν και θα δούμε ότι πάνε προς την ίδια κατεύθυνση όλα. Αν υπήρχε απόκληση, να ξέρετε ούτε άλλες δυνάμεις ήταν απόλυτα συνεπείς με τα μηνύματά τους. Εμείς λοιπόν μιλήσαμε ίσως με πολλές φωνές, αλλά δώσαμε το ίδιο μήνυμα. Στηρίξαμε με όλες αυτές τις προσπάθειες αυτή την αλλαγή η οποία πρέπει να ξεκινήσει τώρα, όπως λέμε. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο πάντως μπορούμε να στηρίξουμε ώστε να υπάρξουν ελεύθερες εκλογές, ορθές εκλογές, αλλά μια δημοκρατία δεν είναι μόνο εκλογές. Είναι και αυτό που λέμε στα αγγλικά institutional building, δηλαδή να ετοιμάσουμε τους θεσμούς, να ετοιμάσουμε τον κόσμο, να ενισχύσει τους θεσμούς έτσι ώστε όσοι θέλουν να στηρίξουν ε, τα δίκαια αιτήματα του λαού να μπορούν να το κάνουν βασιζόμενοι σε μέσα, σε οργάνωση που υπάρχει και έτσι να οδηγηθούν στις εκλογές. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο πρέπει εμείς να φροντίσουμε να ενισχύσουμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις ώστε μαζί να χτίσουν μια νέα και δημοκρατική Αίγυπτο. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο αλλαγών πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Εξού και η δήλωσή μα. Η δήλωσή μα είναι μια κοινή δήλωση των 27 που στέλνει αυτό ακριβώ το ξεκάθαρο μήνυμα στήριξη του Αιγυπτιακού λαού. Έρχομαι τώρα στην ανταγωνιστικότητα και τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Ακόμα και αν κυκλοφόρησαν κάποια χαρτιά, δεν υπάρχει καμία πρόταση, κανένα σχέδιο που να έχει τεθεί στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου. Καμία πρόταση, κανένα μέτρο. Όχι. Μιλάω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε. Εγώ ήμουν εκεί, εσείς δεν ήσασταν εκεί. Λοιπόν, σας λέω, καμία πρόταση δεν τέθηκε. Ούτε από μία, ούτε από δύο χώρες, ούτε από δύο μαζί, καμία. Αυτό που συζητήσαμε είναι τι να κάνουμε. Διότι έχουμε ήδη έναν συντονιστικό μηχανισμό. Έχουμε ένα μηχανισμό σύγκλησης ήδη. Υπάρχουν οι έξι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η έκθεση της Task Force. Οι αποφάσεις που πήραμε ήταν ότι το Μάρτιο σε επίπεδο Συμβουλίου θα έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οικονομική διακυβέρνηση. Όμως υπήρχαν προτάσεις που πηγαίνανε προς την εξής κατεύθυνση. Μήπως θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομική διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ίδιος είπαμε ναι βεβαίως εφόσον και υπάρξουν νέες ιδέες, εφόσον θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση βεβαίως μέσα στην Ευρωζώνη, εφόσον έχουμε κοινωνόμισμα, γιατί όχι, γιατί να το αρνηθούμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε, χωρίς όμως να προκαταλαμβάνει τα πράγματα, χωρίς να υπάρχει κάτι στο χαρτί που να εγκριθεί, ζητήσαμε εγώ ίδιος από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και να έρθουν το Μάρτιο στο Συμβούλιο να μας πούνε. Και σίγουρα και σε κάποιο Συμβούλιο της Ευρωζώνης. Να έρθουν λοιπόν και να μας πούνε τι ακούσανε σε επίπεδο χωρών μελών και τι νομίζουν ότι πρέπει να προτείνουμε. Γιατί και ο κύριος Βαρόσο και εγώ πιστεύουμε ότι πρέπει να τεθούν προτάσεις και όσον αφορά το περιεχόμενο και όσον αφορά τη διαδικασία. Και όσον αφορά το περιεχόμενο και επί της ουσίας και επί του θεσμικού. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Αφού ορισμένοι θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Ξεκινάμε όμως από το μηδέν. Θα γίνουν διαβουλεύσεις από την επόμενη εβδομάδα και θα προτείνουμε μαζί το Μάρτιο κάτι κατά τη διάσκεια του Συμβουλίου της Ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό έγινε. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καλή εξέλιξη, γιατί κύριε Ντόλ, θέλουμε να πάμε προς την κατεύθυνση που είπατε. Περισσότερη Ευρώπη. Βεβαίως. Και γι' αυτό και στο κείμενο λέει σύμφωνα με τις συνθήκες, in line with the treaties. Και γι' αυτό ακριβώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Προεδρία του Συμβουλίου με την Προεδρία της Επιτροπής θα συνεργαστούν, τα θεσμικά όργανα δηλαδή μαζί θα συνεργαστούν για να καταλήξουμε σε προτάσεις όσον αφορά την Ευρωζώνη για να είμαστε περισσότερο συνεκτικοί μεταξύ μας, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην οικονομική μας πολιτική. Για την Αίγυπτο τώρα παρά τις υπερβολικά πολλές φωνές που ακούστηκαν, τελικά περάσαμε ένα και το αυτό μήνυμα. Και αυτό έχει σημασία, ότι είμαστε με τον Αιγυπτιακό λαό κατά τη μεταβατική περίοδο, αυτήν τη τόσο λεπτή και ευαίσθητη που ξεκινάει τώρα. Και ότι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Το μέλλον της Αιγύπτου είναι στα χέρια των ίδιων των Αιγυπτιών, αλλά εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα προχωρήσουμε και για την οικονομική διακυβέρνηση θα υποβάλουμε ένα σχέδιο το Μάρτιο, το οποίο θα ετοιμάσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να έχουμε περισσότερη οικονομική διακυβέρνηση. Δεν είναι κάτι που σας το λέω έτσι τεχνητά και προσπαθώ να δείξω ότι, είναι, ότι είμαι αισιόδοξο. Όχι, η φιλοδοξία υπάρχει. Φάνηκε και τι τελευταίε εβδομάδε και φάνηκε και από τις αγορές, παρόλο που οι αγορέ δεν είναι ο μόνο δείκτη που μα δείχνει αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο φαίνεται να υπάρχει εμπιστοσύνη από τι αγορέ, στα μέτρα, τα τόσο θαραλέα που παίρνουν οι χώρε μέλη και στα σχέδια που έχουμε μέχρι τώρα ετοιμάσει και αυτά που θα ετοιμάσουμε στο μέλλον. Είμαι λοιπόν αισιόδοξο βάσει πεπιθήσεων και αποφάσεων και όχι εξορισμού. Πρόεδρος, θα ξεκινήσει η διαδικασία... Για διαδικαστικό θέλετε το λόγο κύριε Μάλιστα πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτή είναι η διάσκεψη των πρόεδρων. Α? Και ακόμα είμαι πρόεδρος ομάδος μου. Έχω μια ερώτηση λοιπόν προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου για να διευκρινιστεί ένα σημείο. Αυτό το έγγραφο που σας δείχνω λέει σύμφωνο για την ανταγωνιστικότητα. Είπατε ότι αυτό το έγγραφο δεν υπευλήθη στο Συμβούλιο. Σωστά σας κατάλαβα. Το γνωρίζατε πριν από την αρχή της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Το γνωρίζατε. Σας το υπέβαλε η κυρία Καγκελάριος και ο πρόεδρος της Γαλλικής ε, Δημοκρατίας. Ναι. Και γιατί. Εάν δεν το ξέρατε, τι έχετε να πείτε που ο κύριο Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή το υπέβαλαν σε μια ξεχωριστή συνέλευση τύπου. Είδα το έγγραφο. Από όσο ξέρω δεν είναι γαλλογερμανικό αυτό το έγγραφο. Από όσο ξέρω δεν είναι γαλλογερμανικό αυτό το έγγραφο. Και δεύτερον, δεν υπευλήθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν συζητήθηκε εκεί. Και όταν αναφέραμε Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο, αλλά δεν υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Διαδικασία εκτάκτων, εκτάκτων παρεμβάσεων. Μαρία Νταγκράτσια Καρβάλιο, one minute please. Madame Carvalho, one minute please. Moment. Madame Carvalho. Κυρία Καρβάλιο, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρώπη χρειάζεται να ασκήσει πολιτική καθαρής ενέργειας και είμαστε σε καλύτερη θέση για να το κάνουμε αυτό αν συγκρίνουμε με τους ανταγωνιστές μας. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο Βαν Ρομπόη και το Συμβούλιο για την επιλογή να, ε, να, της ενέργειας και της καινοτομίας ως θέματα αλλά λυπάμαι για την φιλοδοξία των συμπερασμάτων, την έλλειψη μάλλον φιλοδοξίας των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και τα συμπεράσματα για την ενέργεια και την καινοτομία θα έπρεπε να είναι ξεχωριστά θέματα. Καινοτομία στην ενέργεια μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη απάντηση για την κρίση σε αυτήν την κρίσιμη φάση όπου αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση μαζί με παγκόσμια ενεργειακή κρίση είναι επίγον να δράσουμε και υπάρχει τρόπος να βγούμε από την κρίση χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε ενέργεια στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ένα λεπτό. Πού είναι ο συνάδελφος Κουμουτσάκος, δεν σας βλέπω. Κύριε Καρβάλιο, πρέπει να κλείσετε το μικρόφωνο σας, μάλλον δεν είναι παρόν. Ο κύριος ε, Γιάσεκ Σάιρους Βόλς και ένα λεπτό. Ε, η ερώτησή μου απευθύνεται στον πρόεδρο Ρομπάι. Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με δύο βασικά θέματα ενέργεια και Μέση Ανατολή Αίγυπτος αλλά τα δύο αυτά θέματα Όλο παραδόξω δεν συνδέθηκαν μεταξύ του. Ποια είναι η εκτίμηση λοιπόν στο Συμβούλιο σε σχέση με τι πιθανέ επιπτώσει τη αλλαγή ε, στην περιοχή όσον αφορά την ίδια την ασφάλεια για την ανεφοδιασμό σε ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επιπτώσεις στην κρίση, ακόμα και αν δηλαδή πραγματοποιηθεί το χειρότερο σενάριο, δηλαδή κλείσει το ιδιόργα του Σουέζ. Ποιες είναι λοιπόν οι οικονομικές ε, και πολιτικές αλλά και ε, επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ κυρία Χέρτζοκ. Σας ευχαριστώ. Για την ενέργεια και το τομέα πιστεύω πως θα είχαμε μπορέσει να πετύχουμε περισσότερο. Τουλάχιστον έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Δυστυχώ, οι πόροι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε να υλοποιηθούν τα προγράμματα αυτά και το Συμβούλιο δεν, έδωσε, δεν συμφώνησε από αυτού. Εγώ πιστεύω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό ωστόσο να έχουμε οικονομική σταθερότητα, άσχετα από το αν μια χώρα ανήκει στην Ευρωζώνη ή όχι. Αν δούμε όμως ε, τις προτεραιότητες της ανταγωνιστικότητας ε, στις, για τις κυβερνήσεις ε, της Ευρωζώνης, θα δούμε ότι βασικά Πολλά λόγια ακούγονται, κυρίως από τη δική μου κυβέρνηση. Πρέπει αυτό να σταματήσει και εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε μεγάλο φόρτο, μεγάλη ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε το θέμα στο μέλλον. κυρία Ελιάνα Γιώτοβα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις αποφάσεις του τελευταίου Συμβουλίου υπογραμμίσατε πολλές φορές ότι η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει την προμήθειά της όσον αφορά την ενέργεια. Δεν πρέπει να, να και μία άλλη στρατηγική για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Συγχρόνως υπογραμμίσατε ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την εταιρική σχέση μας με τη Ρωσία. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποια είναι η γνώμη σας για την δημιουργία του σχεδίου South 3, South Stream, όσον αφορά δηλαδή τα δύο αυτά σχέδια και κυρίως το South Stream. Ποια είναι η γνώμη σας και τον Αμπούκο. Παρακαλώ ένα λεπτό. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούω από την Επιτροπή ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και περισσότερη ανεξαρτησία όσον αφορά την προμήθεια ενέργεια. Νομίζω ότι δεν διαβάζουμε τέτοια πράγματα εκείνο και εγώ. Εγώ το βλέπω ανάποδα. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον προ τα πίσω πάμε. Όταν έχουμε να κάνουμε τώρα και για τις υποδομές για την ενέργεια και εκεί η γλώσσα δεν είναι όπως ήταν πριν, είναι πιο δύναμη προς τα πίσω πάει η Επιτροπή και για αυτό το σχέδιο όσον αφορά τις υποδομές. Αν ήμουν από τις καινούριε χώρες θα ανισχούσα πάρα πολύ για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τέλος, όσον αφορά την χρηματοδότηση της ενέργειας, πουθενά δεν γίνεται μία χρηματοδότηση της ε, τεχνολογίας για την ενέργεια, στρατηγική τεχνολογία. Άρα λοιπόν τίποτα το καινούριο, μάλλον πίσω πάμε παρά μπροστά. Ο κύριος Τρουν Στίβενσον τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ενθουσιάστηκα που άκουσα τον Πρόεδρο Φανορομπάη να λέει ότι θα στηρίξουμε το λαό της Αιγύπτου. Ω προς αυτό ο Γκραντά είπε στον Αλχαμανή του Ιράν ότι θα στηρίξει τον λαό της Αιγύπτου. Καλή παρέα έχουμε, όπως στηρίζει και το λαό της Τινησίας στη δική του εξέγερση και της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ ε, κατέπνιξε την ε, εξέγερση στο Ιράν και μόλις θα τον περασμένη μόλις εβδομάδα έναν Ολλανδό ε, ε, ε φυλάκισαν γιατί διαμαρτυρήθηκε κατά του Αχμαντίνη Λοιπόν, ε, οι Ολλανδοί διαμαρτυρήθηκαν. Εμεί τι κάνουμε για να στηρίξουμε το λαό του Ιράν. Αφήστε το λαό τη Αιγύπτου. Μα στηρίξτε το λαό του Ιράν κατά του πιο φασιστικού και καταπιστικού καθεστώτος στον κόσμο. Ευχαριστώ, κύριο Στούσα. Η αποκωδικοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τα μέσα και οι αποφάσει του σηματοδοτούν νέα δεινά για του λαού. Σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε το κείμενο που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής δεν είναι στα γαλλικά, είναι στα γερμανικά. Αλλά αποτελεί πρόταση και σας ρωτώ συγκεκριμένα. Πρώτο ζήτημα. Τέθηκε θέμα στο Συμβούλιο τα έξι σημεία ως εξής. Πρώτο, κατάργηση των συστημάτων αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών των εργαζομένων. Δεύτερο, διεύρυνση και επιτάχυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πτυχίων για την προώθηση της κινητικότητας των εργαζόμενων στην Ευρώπη. Τρίτο, προσπάθεια για τη δημιουργία ενιαίας βάσης υπολογισμού του φόρου των επιχειρήσεων. Τέταρτο, προσαρμογή του συνταξιοδοτικού συστήματος στη δημογραφική ανάπτυξη, σύνδεσή του με το προσδόκιμο ζωής. Πέμπτο, υποχρέωση για φρενάρισμα του χρέους στα συντάγματα όλων των κρατών μελών ανάλογα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έκτο εισαγωγή μέτρων σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ. Ε, Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα μέτρα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης αποτελούν ένα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αλλά υπάρχει μια συμφωνία για τον ανταγωνισμό και σε άλλους τομείς όπου οι χώρες μας βρίσκονται πιο πίσω. Ένας τέτοιος τομέας είναι οι πληρωμές που γίνονται για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων που έχουμε από την καινοτομία. Για συγκρίνετε τι γίνεται με την Κίνα. Στην Κίνα, άμα θέλουν να λύσουν ένα πρόβλημα, αντιγράφουν απλώς και μόνο και χωρίς καμία διατύπωση προωθούν μετά την ιδέα του στον κόσμο. Ενώ εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατεύουμε την ε, πατέντα, την πνευματική ιδιοκτησία κλπ αλλά έτσι μένουμε πίσω. Θα έπρεπε να απλοποιήσουμε λοιπόν τις διαδικασίες για να τα καταφέρουμε. Ένα άλλος, τομέα τομέας είναι οι δυσκολίες που βάζουμε και τους επιχειρηματίες. Ένας ε, φούρναρης ή ένας εστιατόρας πρέπει σε έξι ε, οργανισμούς στη χώρα μου να δίνουν στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο επίσημο ημερησία διάταξη υπήρχε το θέμα ενέργεια. Όλοι όμω μιλάνε για το σύμφωνο της αγωνιστικότητας. Σας ρωτώ λοιπόν, πού είναι η επικοινωνία, η διαφάνεια. Και δεύτερον θα ήθελα σύντομα να πω το εξής. Η διεύρυνση ε, των μέτρων ε, ασφαλείας θα, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν μπορεί να μείνει εκτός νυφών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς έχετε κατά νου λοιπόν να εμπλακεί η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαζινιώρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στη νότια όθη της Μεσογείου οφείλεται και στα δικά μας φάλματα, στην ε, ανικανότητά μας να καταλάβουμε τα όσα ποάζονταν στους λαούς αυτών των χωρών. Έπρεπε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μέσω ε, ισχυρών θεσμικών ε, οργάνων. Σήμερα πληρώνουμε την ανεπαρκή ανάπτυξη σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Πρέπει να διαπιστώσουμε την αποτυχία τη διαδικασία τη Λισαβάνης, της, της, ε, Βαρκελόνης, συγγνώμη, επίσης την αποτυχία τη Ένωση για την Μεσόγειο, αλλά και την ανεπάρκεια τη Ευρωπαϊκή στήριξη, αλλά και την ανεπάρκεια τη δική μα δομή, Και εδώ αναφέρομαι στην Υπηρεσία εξωτερική δράση που απέδειξε ότι δεν ξέρει να προβλέπει, ούτε και να ε, καλύπτει τις ε, θέσεις. Πρέπει λοιπόν να, ε, να ρωτήσω στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο αν και πώς σκοπεύουν να προωθήσουν σημαντικά προγράμματα για την ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρηματικού ιστού των χωρών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. συνάδελφος Ζαμπιέρ Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μια κλασική κατάσταση. Ο Σούλς που επικρίνει την Μέρκελ και ο Φερχόφστατ που επικρίνει τον Σαρκοζή επικρίνουν την διακυβερνητικότητα. Αναφέρατε, κύριε Φερχόφιστα, δύο παραδείγματα. Στρατηγική Λισαβόνα και Σύμφωνο Σταθερότητα. Αλλά για τη στρατηγική τη Λισαβόνα, εγώ εξελέγει το 2005. Η Κομισιόν μα ειδοποίησε για το γεγονό ότι πηγαίναμε ε, προ την αποτυχία. 21 διαδικασίε παραβίαση για το Σύμφωνο Σταθερότητα το Σεπτέμβριο του 2008. Δεν μπορούσε να έχει ξεκινήσει διαδικασίε επιπαραβίαση νωρίτερα η Κομισιόν. Η Κομισιόν πρέπει να ειδοποιεί εγώ πιστεύω πως στην πράξη είμαστε συνυπεύθυνοι για μια κατάσταση και σήμερα ας μην επικρίνουμε τους επικεφαλείς κρατών που κάνουν ό,τι μπορούν και είναι Ευρωπαίοι. Ε, σήμερα θα πρέπει από κοινού να προχωρήσουμε, πράγμα που με οδηγεί κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, να σας ζητήσω να έχετε με το Κοινοβούλιο μας πιο ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς. Όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σα, σα είχα προτείνει να έρθετε αμέσω ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έγινε αυτό όμω και πιστεύω πως ήρθε η ώρα πια να έχετε περισσότερους δεσμούς μαζί μας και συζητήσεις μαζί μας. Σας ευχαριστώ, Διακόπτη. Ο Πρόεδρος, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Καλφίν. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φανρόπαη, θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ μαζί σας ε, όταν λέτε ότι δεν προτείνετε καμία αλλαγή η οποία θα επέτρεπε να περάσουμε στην κοινοτική μέθοδο. Αυτό γίνεται με συνεπλές συνθήκες Λισαβόνας. Υπάρχει ο, αυτή τη στιγμή μία στροφή προς την διακυβερνητική μέθοδο. Όλα αυτά που συζητάμε μέσα στον χώρο του Ευρωζώνης οδηγούν σε μία διάσπαση μεταξύ των χωρών ευρώ και των μη χωρών ευρώ. Εσείς ως πρόεδρος του Συμβουλίου τι συστήνετε να ψηφίσει το Συμβούλιο για να μπορέσει να προωθήσει την κοινοτική μέθοδο για να μην υπάρχουν ε, διάφοροι αποκλειστικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούν όλες οι χώρες να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σαλβάρο Αλεξάνδερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια υποσημείωση για την Αίγυπτο. Το αποτέλεσμα της κακοφωνίας στην ευρωτονική πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Ευρώπη ήταν η δημιουργία της, ε, της θέσης της ε, υπηρεσίας πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής δεν επιτρέπεται πάλι να σιωπούνε ε, γιατί για την αιτή σιώπησε η κυρία Άστον, για την Αίγυπτο σιώπησε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζα, αλλά θα πρέπει να μπορεί να ακουστεί, να υψώσει τη φωνή της και να ακούγεται. Η κυρία Αστον, όσον αφορά το σύμφωνο του ανταγωνισμού, είπατε τι έγινε στο Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να είναι ανησυχητικό ότι και η Γαλλία και η Γερμανία προσπαθούν εκτός των θεσμικών οργάνων να προχωρήσουν και να μην τα βάλουν αυτά στις θεσμικά όργανα και στη θεσμική διαδικασία. Ρωτώ λοιπόν, εσείς μπορείτε να μας πείτε ότι ερκίζεστε στην κοινοτική διαδικασία ή προτιμάτε τη διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊ... ε, όπως υπάρχει μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και τελειώνω το γεγονός ε, ότι πρόκειται να συνεργαστούν τα κοινοβούλια της ζώνης ευρώ θα δημιουργήσει ένα νέο, ε, ένα νέο κοινοβούλιο. Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τόσα έχουν γίνει στην Αίγυπτο. Μην ξεχνάμε και την επίθεση που έγινε με τους Κόπτες, τους κόπτες. Συνεχίζουν να καίγουν εκκλησίες. Και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και αλλού. Κύριε Φαναραμπάου, γιατί στα συμπεράσματά του για την Αίγυπτο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ανέφερε τίποτα όσον αφορά τους κόπτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει εδώ η ομιλία μα 14 συνάδελφοι, 14 μίλησαν. Με συγχωρείτε που δεν μπορούσαν να μιλήσουν όλοι. Ακολούθησα τον κατάλογο που είχα μπροστά μου. Σε βάση την σειρά με την οποία είχαν γραφεί. Ο αντιπρόεδρο Σέκτοβης έχει uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε πραγματικά περισσότερη Ευρώπη, όπω είπε και ο κ. Ντόλ, και το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στον τομέα τη ενέργεια. Και εμεί στην Κομισιόν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε πολύ ε, ξεκάθαρε προθυμίε, δηλαδή μέχρι το 2014 θα πρέπει να έχουμε εσωτερική αγορά για την ενέργεια, το 2015-2016 θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις τελευταίες νησίδες ενέργειας στην Ευρώπη και σας διαβεβαιώ όταν πρόκειται για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα θα προχωρήσει η Κομισιόν και δεν εφαρμοστεί σωστά το κοινοτικό και εκτιμένο στις εθνικές νομοθεσίες εμείς θα προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτά που μας επιτρέπει η συνθήκη γιατί ξέρουμε ποια θα είναι το όφελος για την Ευρώπη ποιο θα είναι το όφελος για τον Ευρωπαίο πολίτη εάν έχουμε τελικά καλά λειτουργούσε η εσωτερική αγορά στον τομέα της ενέργειας. Το ίδιο θα μπορούσα να πω για τον τόσο σημαντικό τομέα της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας όπου ελέγχθη επίσης. Εδώ θα πρέπει πραγματικά να εκτιμήσουμε την ειλικρίνεια των συμπερασμάτων που λένε ξεκάθαρα έχουμε καθυστέρηση σε αυτό τον τομέα. Στην αποτελεσματική χρήση δηλαδή της ενέργειας και βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Και η Κομισιόν είπε ξεκάθαρα ότι εάν δεν υπάρχει θετική εξέλιξη μέχρι το 2013 θα αναλύσουμε προσεκτικά την κατάσταση και αν χρειάζεται θα προχωρήσουμε σε προτάσεις για νομικά δεσμευτικούς στόχους. Έχουμε δυνατότητες εφαρμογής σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ για τα συμπεράσματα αυτά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο σημείωσε ότι η η ενεργειακή πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική για κάθε κράτος μέλος, για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θέλουν να προχωρήσουν πραγματικά αποτελεσματικά για να δημιουργήσουν την εσωτερική αγορά και να ενδυναμώσουν την ασφάλεια τροφοδότηση της ενέργειας, όπως είπε και ο κ. Σαρισβόλσκι. Όσον αφορά την ασφαλή τροφοδότηση, θα πρέπει να εξάσουμε και τι δύο πτυχέ. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια αυτή, βελτιώνοντα τι εσωτερικέ κοινωτικέ πολιτικέ. Το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις και οι μηχανισμοί της αγοράς που εργάζονται στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις εκδοτικέ μας πολιτικές όταν πρόκειται για επικοινωνία με τους εταίρους μας, με εκείνους που μας προσφέρουν τις ε, πηγές αυτές της ενέργειας, πώς θα μπορούμε να προβλέπουμε τα ενδυνάμει προβλήματα των περιοχών από τι οποίες παίρνουμε την ενέργεια και θα μπορέσουμε νομίζω να καθαρίσουμε απόλυτα σαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε για εκείνους που προ... μας προμηθεύουν την ενέργεια για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την συνεργασία. Γι' αυτό η αναφορά στο South Stream ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει πραγματικά να ενδυναμώσουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να ανοίξουμε νέες πηγές ενέργειας για την Ευρώπη. Περνώντα στην ε, οικονομική διακυβέρνηση, εδώ θα πρέπει νομίζω να εκτιμήσουμε την πρόοδο που πετύχαμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Εάν, δεν, εάν υπήρχε ένα θετικό στοιχείο στην οικονομική κρίση, ήταν ακριβώ ότι αναγνωρίσαμε πώ είμαστε αλληλοσυνδεδεμένοι, ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μα, να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και νομίζω ότι πετύχαμε πρόοδο. Εάν πριν από δύο-τρία χρόνια είχαμε αναφέρει ότι θα είχαμε μια τέτοια συζήτηση για τους εθνικούς προπολογισμού εδώ στην Ευρώπη, αυτό θα θεωρείτε ότι ήταν κάτι που θα γίνει ίσως κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Δεν θέλω να αναφερθώ και στα μέτρα μεταρρύθμιση ε, για τα οποία η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη που προσπαθούμε να τα ενθαρρύνουμε και να τα να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξου στόχου και πιο σαφεί στρατηγικέ για το μέλλον. Προφανώ λοιπόν αυτά που έχουν γίνει δεν είναι αρκετά. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω και γι' αυτό η Κομισιόν καλασορίζει κάθε προσπάθεια για πιο στενή οικονομική συνεργασία, πιο στενή οικονομική διακυβέρνηση. Οπωσδήποτε υποστηρίζουμε την πρόθεση των κρονών των μελών να συνεργαστούν και στους νέους τομείς. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς τους νέους τομείς βρίσκονται κάτω από το καθεστώς των εθνικών δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να ασπαστούμε όποια μορφή οικονομικής διακυβέρνησης προωθεί τους κοινοτικούς στόχους, στην εσωτερική αγορά και θα βασίζεται στην καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη. Και θα πρέπει πραγματικά να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο πρόεδρος των Ρομπόη. Ότι ούτε η Κομισιόν είχε πάρει κανένα γάλλο-γερμανικό μη έγγραφο και οπωσδήποτε δεν συζήτησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και γι' αυτό η απόφαση που ελήφθη είναι ότι θα έχουμε πάρα πολύ στενές διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της Ευρώπης για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις πολύπλοκες λύσεις, πολύπλοκη προσέγγιση για τη διάσκεψη προφή του Μαρτίου. Τέλο για την Αίγυπτο και την Ισία. Προφανώ και στι δύο χώρε η κατάσταση είναι πολύπλοκη και η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων συνεργάζονται για να μπορέσουν να δουν πώ θα μπορέσουν καλύτερα να εκμεταλλευτούν τι δυνατότητε που έχουμε στη διάθεσή μα για να υποστηριχθεί η μετάβαση στη δημοκρατία, στη δημοκρατία συγγνώμη, των χωρών αυτών και να δούμε πώ θα τους ε, παρουσιάσουμε τις καλές πρακτικές και πώς θα ε, ε, δημιουργηθεί έτσι η δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι πριν την προηγούμενη φορά είχα μιλήσει πάρα πολύ. Οπότε φτάνει, Πρόεδρε. Σωστά. Το λέει για όλους, λέει ο κύριος Φερχόφστατ από την αίθουσα. Για το Ιράν, λέει ο πρόεδρος Φαν αξιότιμοι συνάδελφοι, Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε επιπλέον κυρώσεις εξαιτία των ε, πυρηνικών πρωτοβουλειών του Ιράν. Κυρώσεις οι οποίες για πρώτη φορά είχαν επιπτώσεις και έφεραν το Ιράν εκ νέου στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, για το Ιράν έχουμε μία σαφή θέση. Και συγχρόνως πολύ σκληρή αλλά αποτελεσματική. Εξάλλου η ίδια η κυρία Άστον είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων που γίνονται με το Ιράν ως επικεφαλής των έξι χωρών που διαπραγματεύονται με το Ιράν. Άρα είμαστε ιδιαίτερα παρόντες στο ιρανικό ζήτημα και αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας. Για το θέμα του ανταγωνισμού. Πολλοί από εσά είπαν ότι υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός και εξωτερικός ανταγωνισμός. Για τον εσωτερικό θα κάνουμε πολλά ε, μετά από την έκθεση της Task Force και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά συγχρόνως πρέπει να φροντίσουμε για τη στρατηγική 2020. Να έχουμε δηλαδή και σε παγκόσμιο επίπεδο ε, γερή θέση να είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί τελειώ δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιος από εσά είπε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να συζητήσουμε τις νέες προτάσεις για την διακυβέρνηση μετά από την έκθεση που θα ετοιμάσουμε ο κύριος Μπαρόσο και εγώ. Ενδιαφέρουσα πρόταση να το συζητήσουμε με τον πρόεδρο Πούτσεκ και σίγουρα στη διάσκεψη των πρόεδρων θα δούμε πόσο στο δεύτερο δεκαπεθήμερο του Μαρτίου θα μπορέσουμε να έχουμε και το Κοινοβούλιο μαζί μας προκειμένου να καταλήξουμε στις τελικές προτάσεις. Τώρα, για την Ευρωζώνη και τους άλλους. Στην απόφαση ακριβώς είπαμε ότι αυτοί που δεν είναι μέλη στην Ευρωζώνη πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην οικονομική διακυβέρνηση. Αν διαβάσετε προσεκτικά τα αποτελέσματα θα δείτε και τα συμπεράσματά μας, θα δείτε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε διαβούλευση και να συμμετάσχουν στον οικονομικό συντονισμό. Φυσικά υπό κάποιους όρους. Έχω δύο ακόμα παρατηρήσεις. Και αυτούς που λένε ορκίζεστε στην κοινοτική μέθοδο εδώ. Εγώ μόνο στη συνθήκη ορκίζομαι. Στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και ακριβώς στα συμπεράσματα είπαμε ότι θα δουλέψουμε σύμφωνα με τη συνθήκη. Κάτι το οποίο κάναμε και καθόλου τη διάρκεια της κρίσης στην Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν εγώ τηρώ τις συνθήκες και πάντα τις συνθήκες. Για τις μειονότητες τώρα στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο που στο κείμενο της δήλωσης δύο φορές αναφέρεται ο πλουραλισμός. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία μόνο με την μειοψηφία, πρέπει να σεβόμαστε και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και αυτό εκφράζεται με τη λέξη πλουραλισμός. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ, επικεφαλής πολιτικών ομάδων και τους υπόλοιπους. Έλξη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.